Um, ich darf die Sitzung eröffnen. Ich, uh, frage, ob zur Tagesordnung... Σα ερωτώ για την ημερήσια διάταξη υπάρχουν παρατηρήσει, δεν υπάρχουν. Ο πρόεδρο δεν έχει ανακοινώσει. Και έτσι περνάμε αμέσως στο σημείο 3. Έλεγχη και εφαρμογή ελέγχων όσον αφορά βάσεις δεδομένων για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Έχουμε τις τροπολογίες λοιπόν που εξετάστηκαν από τη νομική υπηρεσία ως ήθιστε και μας είπαν, μας γνωστοποίησαν ότι κάποιες από τις τροπολογίες που κατέθεσε ο κύριος Σαφάουζερ δεν μπορούν να τεθούν σε ψηφοφορία επειδή ξεπερνούν τα εσκαμένα της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Για παράδειγμα η νομική βάση αναφέρεται σε σχέση με τη συνθήκη και διαγράφεται και προστίθεται μια νομική βάση από την ε, δήλωση ε, για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Χαίρομαι όταν υπάρχει η αναφορά στα, στην ε, διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά δεν είναι νομική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νομική βάση. Γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι με βάση αυτές τις ανακοινώσεις και μετά από εξέταση και από εμένα τον ίδιο θεωρούμε και εμείς αυτό ότι δηλαδή οι τροπολογίες 84, 75, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 για αυτό τον λόγο δεν μπορούν να γίνουν δεκτές και δεν θα ψηφιστούν. Για τις άλλες τροπολογίες του κυρίου Σαφάζο φυσικά αυτές θα τις ψηφίσουμε τις άλλες. Υπάρχει αντίρρηση, δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν αποφασίζεται και κυρώνεται. Και περνάμε τώρα στην κανονική διαδικασία ψηφοφορία, ψήφισης. Θα ήθελα ο κύριος Τένοκ όμως πρώτα να μας υποβάλει μια πρόταση που έχει για την ψηφοφορία ή πώς έχει αυτό. Παρακαλώ κύριε Τένοκ. Κάτι διαφορετικό θέλω να πω, Πρόεδρε, ότι έχουμε ε, συνολική ψηφοφορία, unblock, για την έκθεση όσον αφορά τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα. Υπάρχουν όλες τροπολογίες αφαόρ, οι μεγάλες ομάδες είναι κατά, οπότε αν τις ψηφίσαμε όλες μαζί θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Πρόεδρος. Δεν είναι μια ανελακτική, αλλά πρόσθετη η πρόταση. Ένα μέρος των τροπολογιών έχει ήδη διαθετηθεί. Οι άλλες τροπολογίες μπορούν ε, ομού να ψηφιστούν. Υπάρχει κάποια αντίρρηση να μην γίνει αυτό. Δεν υπάρχει. Εντάξει, τότε λοιπόν. Παρακαλώ εσείς, τι λέτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι τροπολογίες πρέπει να ψηφιστούν όχι αλλά μία-μία χωριστά διότι κάθε μία από αυτές έχει και την σημασία της και την έννοιά της. Υπ' αυτή την έννοια δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα ψηφίσουμε συνολικά αντροπολογίες χωρίς να τις εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Ε, επαναλαμβάνω και αργά για να προλαβαίνει η μεταφραστική υπηρεσία να μεταφράζει. Δεν συμφωνώ με την πρόταση. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε συλλήβδιν χωρίς να εξετάσουμε τις ε, τροπολογίες. Κάθε τροπολογία έχει τη δική της έννοια και αναφέρεται σε συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα βάλουμε όλα σε ένα καλάθι και να τα ψηφίσουμε όλα μαζί. Δεν συμφωνώ με αυτή την πρόταση. Stimmen. Λοιπόν, για αυτές τις τροπολογίες, ε, για το, την απόφαση που θα ληφθεί τώρα ψηφίζοντας, ποιοι είναι υπέρ του ομού να ψηφιστούν οι τροπολογίες αυτές της Σαφχάουζερ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν. Λοιπόν αποφασίστηκε και εγκρίθηκε. Γι' αυτό παρακαλώ τώρα πρώτα-πρώτα να το κάνουμε αυτό. Ποιοι είναι υπέρ των τροπολογιών Σαφχάουζερ, να σηκώσουν το χέρι υπέρ κατά αποχές Απορρίφθηκαν λοιπόν ομού οι τροπολογίε Σαφάουζερ. Περνάμε στην τροπολογία 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 79 υπέρ. Κατά αποχές και πάλι 79 υπέρ κατά έλεγχος θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρχεται ψηφίζουμε την 79 Εντάξει. That's your problem. Δικό σας πρόβλημα αυτό. Αν είναι πολύ μικρή η διαφορά, τότε να μας το υπενθυμίσετε, εντάξει. Okay. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας, λοιπόν. Απορρίφθηκε. 21, 21 υπέρ, 36 εναντίον. Απορρίφθηκε. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 80 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 81 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 84 λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Βεργιά από την 22 27 ομού συνολικά μπορούμε να τις ψηφίσουμε όχι λέτε 22 υπέρ, λοιπόν, 22 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 24 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 25 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε λοιπόν, ψηφίζουμε την 25, άρχεται. It's closed. Πέρας ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα έγινε δεκτή. 32 υπέρ, 27 εναντίον. Με μία αποχή. Λοιπόν, 26 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 30 υπέρ. Schaffhauser. Ταυτόσημη και έτσι καταψηφίστηκε, καταπίπτει η Schaffhauser. Τροπολογία 30 λοιπόν, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Καταπίπτει αυτή η 3 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 40 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 41 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 42 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 45 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 46 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 47 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 51 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 52 υπέρ. 55 συγγνώμη υπέρ. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Υπέρ της γνωμοδότησης τώρα συνολικά ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε άρχεται. And Das hmm? Ergebnis ist Εγκρίθηκε η έκθεση με 54 υπέρ, 8 εναντίον και α, αποχή. Είχα και εγώ συμμετάσχει. Εντάξει, ευχαριστώ. Για να προσέχετε το λέω. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην έκθεση για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, εισηγητή ο κύριος Νάρτ. Ο κύριος εισηγητή θα ήθελε να κάνει κάποια παρατήρηση. Όχι. Ξεκινάμε αμέσως με την ψηφοφόρη, με την ψήφιση. Τροπολογία 71, υπέρ. Κατά. απόχέ. Απορρίφθηκε. 11, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 100 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 102 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 101 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 104 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 103 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβαστική 4 συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πάμε τώρα στην τροπολογία 108 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 109 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 110 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 111 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 112 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 113 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 114 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 118 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 119 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Για την 119 έλεγχο. Αυτό ζητήσατε. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας με 30 υπέρ και 31 εναντίον απορρίφθηκε 31 εναντίον 30 υπέρ απορρίφθηκε 31 εναντίον 30 υπέρ απορρίφθηκε τι να κάνουμε κοιτάξτε λοιπόν τους αριθμούς μετρήσαμε και ένας ήταν εναντίον απορρίφθηκε λοιπόν καλή προσπάθεια κύριε Φανόρδεν συνεχίζουμε Λοιπόν, ποια ήταν αυτή η 119 119 υπέρ, λέει ο πρόεδρος. Αυτή ήταν η 119 που ψηφίσαμε, ωραία, η 120 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 100... Έλεγχος, η 120. Ψηφίζουμε την 120 ηλεκτρονικά, άρχεται. Αλλά, der Freund gibt mir ein Whisky aus. Ο κύριος Φρόιντ μετά θα κεράσει ένα ουίσκι, εντάξει. Με 31 ψήφους, 31 υπέρ, 30 εναντίον εγκρίθηκε. Εντάξει, θα το κεράσω εγώ. Περνάμε στην τροπολογία 16 και 122 υπέρ αυτών. Κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίζουμε την 16 και 122 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Θα είναι πολύ δαπανηρό λοιπόν. Πέρα ψηφοφορία με 32 ψήφου υπέρ 27 εναντίον εγκρίθηκαν. Περνάμε στο συμβιβασμό 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 126 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 127 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 128 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 18-129 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν 130 ναι ήταν σαφές όμως το αποτέλεσμα οι σοσιαλιστές ψήφισαν με διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά τι να κάνουμε 130 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 131-132 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν 133 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 19 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίζουμε την 19 άρχεται 19 ελέγχουμε πέρας ψηφοφορίας 34 υπέρ 25 εναντίον με μία αποχή εγκρίθηκε Περνάμε στην 134 υπέρ κατά έλεγχος. Ψηφίζουμε την 134. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 34 εναντίον 25 υπέρ. 135-136 τώρα υπέρ αυτών. Κατά. Αποχές απορρίφθηκαν. Λοιπόν, σκοτσέζικο ουίσκι θα είναι κύριε Τένο, έτσι. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ 42 εναντίον. Απορρίφθηκαν. Περνάμε τώρα στις τροπολογίες που βρισκόμασταν πριν. Ένα λεπτό. Μισό λεπτό. 20, 137 τώρα. Υπέρ αυτών. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. 138 υπέρ, κατά. 138 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 139 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 140 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε 141 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 143 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 21 145 υπέρ αυτών κατά αποχές θα ελέγξουμε 21 145 ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκαν με 33 ψήφου υπέρ 27 εναντίον. Εγκρίθηκαν. Πάμε στην τροπολογία 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 147 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 24-148 υπέρ αυτών. Κατά αποχές εγκρίθηκαν 149-150 υπέρ αυτών. Κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίζουμε 149-150 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκαν 151 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίζουμε την 151 ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε 152 υπέρ κατά αποχές 25153 υπέρ αυτών κατά αποχές 26154 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκαν. Συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 157 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίζουμε την 157 άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Ισοψηφία και απορρίφθηκε. Μια ο ένας, μια ο άλλος. Κοιτάξτε λοιπόν. Κανείς, κανείς δεν το... Δεν μπορώ πέντε να τους μετράω χωρίς να έχουν την κάρτα και να συμμετέχουν. Εντάξει, ας τα επαναλάβουμε λοιπόν. Αν δεν δούλεψε η συσκευή, έστω λοιπόν. Επαναλαμβάνουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 27 υπέρ 31 εναντίον απορρίφθηκε. Αυτή ήταν ε, τούτη εδώ η τροπολογία, έτσι. Ωραία. 158 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 28, 159 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκαν. Συμβιβασμός 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 164 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε 166 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 165 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 167 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 31, 169 και 170 ταυτόσημες υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν Συμβιβασμός 9 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίθηκε. Τροπολογία 174 υπέρ. Κατά απόχέ απορρίφθηκε. 175 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίζουμε την 175 άρχεται. Πέρας ψηφοφορία. 31 εναντίον 23 υπέρ απορρίφθηκε. 176 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Μην το προσπαθείς κάθε φορά. Γίνεται βαρετό στο τέλος τέλος. Ποια ήταν τώρα η 176 ήταν. Πέρας ψηφοφορίας. Κάτι όμως δεν πάει καλά εδώ. Κάτι πήγε στραβά με τέτοιο αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 176 άρχεται. Δεν είναι εδώ έλεγχος συνόρων, είναι έλεγχος ψηφοφορίας. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας. 32 υπέρ 29 εναντίον, μία αποχή εγκρίθηκε. Μάλιστα. 177 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 178 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 180 υπέρ. Κατά αποχές. Και άλλη μία φορά. Ελέγχουμε λοιπόν. 180 άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Okay. I need a... Uh, λοιπόν, εσείς κύριε Πρεκοβίτς θα παναλάβετε την Προεδρία πρέπει να αποχωρήσω αμέσως γιατί διαφορετικά δεν θα προλάβω το αεροπλάνο μου. Και γι' αυτό ο κύριος Πλέγκοβιτς θα προεδρεύσει. Παρακαλώ. True, Καλημέρα. Συνεχίζουμε λοιπόν. 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Νομίζω ότι όλες οι τροπολογίες ε, Σακοράφα έχουν την τύχη των Σαφχάουζερ. Όλοι είναι κατά. Δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε όπως τις τροπολογίες ε, ε, Σαφχάουζεν. Σακοράφα. Γιατί είναι πολλές οι τροπολογίες Σακοράφα. Τέσσερις σελίδες έχουν μείνει για να μην μπερδέψουμε το σύστημα. Ας προχωρήσουμε. it's a lot of pages. It's pages. Okay, then let's try to Uh, Τέλο πάντων, να ψηφίσουμε την πρόταση του κυρίου Γκάλερα. Εγώ δεν έχω το κατάλογο ψηφοφοριών όλων των ομάδων, ε, οπότε αυτό είναι δική σας ε, εντύπωση, εσείς το λέτε αυτό. Υπάρχει μια δουλειά που κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα την απορρίπτουν εκ των προτέρων. Κάναμε τροπολογίες, είμαστε εδώ για να ψηφίσουμε και θα ψηφιστούν με τη σειρά τους. We will continue the vote as it was. Όχι, θα συνεχίσουμε την ψηφοφορία κανονικά. Okay. Χωρίς μικρόφωνο. Okay. Hello. We will continue the vote as it... Συνεχίζουμε κανονικά την ψηφοφορία. Την ψηφίσαμε την 179 νομίζω, έτσι δεν είναι. 33-181 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 34-183 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ κατά αποχές δεκτή 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 Α, 190 ψηφίζουν ηλεκτρονικά 1, 9, 0. Τροπολογία 190. Ψηφίζουμε. Close the vote. Πέρας. Αυτή εγκρίθηκε. Ε, δεν φαινόταν. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν, δεν σηκώνετε τα χέρια σωστά. 192. Ηλεκτρονική ψηφοφορία θα γίνει.

κατά αποχές έλεγχος γιατί μου φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά Ελέγχο, ψηφίζουμε την 194 ηλεκτρονικά πέρας 32 προς 27 Τώρα πάμε στην 195 υπέρ. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 198 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 200 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Έλεγχος γιατί είναι λίγο διαφοροποιημένη η εκλογική σας συμπεριφορά. Ψηφίζουμε τη 200. Πέρας. Όχι, 25 προς 32 απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται 201 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι απορρίπτεται αλλά πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά πέρας 23 προς 36 απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν σηκώνεται τα χέρια όπως πρέπει, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 202. Πέρας. 25 προς 34 απορρίπτεται. 39 κάθετος 203. Νάρτ Κεφαλογιάννης υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 207 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 208 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 209 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42-11-212 2 πέρα. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρας. 33 ε, προς 25 εγκρίνεται. 213 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 214 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά πέρας απερίφθη 22 προς 36 215 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 218 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή 219 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 220 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.23 υπέρ κατά αποχές δεκτεί 2.24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 227 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίζουμε τη 227 ηλεκτρονικά 227 Πέρας. 23 προς 34 απορρίπτεται. 2.28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.32 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. 2.32 ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. 2.32 Λείπουν κάποιοι. Ε, πέρας. Λοιπόν, 29 προς 28. Εγκρίνεται. 2.33 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.36 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.34 υπέρ. Κατά. Κάποιοι ψηφίζουν και τα δύο. Έλεγχος ηλεκτρονικός. 2.34. 2.34 λοιπόν του κυρίου Βαν Όρντεν. Πέρας. Μα, εντυπωσιακό. 13 υπέρ και 45 κατά. Δεν φαινόταν. 43, 2.35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 2.37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.42 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.43 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.44 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 2.44. Πέρας. 23 προς 35 απορρίπτεται. 2.45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο, νομίζω ότι ήταν σαφές όμως. Αν θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίζουμε. Ωραία, ψηφίζουμε τη 245 ηλεκτρονικά. Απερίφθη 23 προς 36. 2.46 υπέρ. Κατά αποχέσε, δεκτή. 2.47 υπέρ. Κατά αποχέσε, δεκτή. 2.48 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.49 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.50 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίζουμε τη 2.50 ηλεκτρονικά 29 προς 29 αυτό σημαίνει ψήφισε κανείς χωρίς κάρτα ψήφισε κανείς υπέρ... Α, α, 30 προς 29 ψήφισε ε, μία συνάδελφος χωρίς κάρτα, άρα πέρασε. Εγκρίνεται. 45-251 ε, υπέρ, κατά. Ποιος είναι κατά του 45-251? Απορρίπτονται. 252 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 253 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 έχει αποσυρθεί. 2.54 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.55 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 256 υπέρ. Κατά. Εκτός μικροφώνου παρέμβαση. Με αγγλικά, για να με καταλαβαίνετε πιο εύκολα, λέει ο πρόεδρος. Εκτός μικροφώνου παρέμβαση από την αίθουσα, δεν την ακούμε. Δεν κατάλαβα και εγώ τι έγινε. Α, στα αγγλικά τα νούμερα δεν τα λέω καλά. Λοιπόν, 256 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 261 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 48 κάθετος 263 υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 48-263 ψηφίστε παρακαλώ. πέρα τη ψηφοφορια 33 33-25 υπέρ, εγκρίνεται δηλαδή. 262 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 262, ψηφίστε. Άλλοι δύο-τρει να ψηφίσουν παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. 22-35. Απορρίφθηκε. ...264 υπέρ, κατά, αποχές. Ωραία, θα ελέγξουμε. 264. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται 35-22. 49. Υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει, συγγνώμη. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 267. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι σοσιαλιστές είναι υπέρ ή κατά, ρωτάει ο πρόεδρος. Εγκρίθηκε τότε. 267 να ελέγξουμε, ωραία. 267 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πολύ διχασμένοι οι σοσιαλιστές. Λοιπόν, 267 πέρα της ψηφοφορίας. 24-35 το αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 268 υπέρ. Το ΕΛΚ είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 269 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 270 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 271 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 272 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 273 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 274 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 275 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 276 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 277 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 278 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 279 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 280 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 281 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 56-282 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 283 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 284 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 285 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 286 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 287 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήταν σαφές το αποτέλεσμα, λέει ο Πρόεδρος. 288 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε αυτήν την 288. Ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ. Άλλοι δύο-τρει να ψηφίσουν. Πέρα τη ψηφοφορία. 31 ψήφοι υπέρ, 25 κατά. 289 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 290 υπέρ, κατά, αποχές, υπέρ. Νομίζω όλα θα ελέγξουμε. 290 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. 30 ψήφοι υπέρ, 25 κατά. 291 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε για τη 291. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. 23 υπέρ, 33 κατά, απορρίφθηκε. 292 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 293 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. 293. Πέρας της φοφορίας. 24 υπέρ 34 κατά απορρίφθηκε. 294 υπέρ. Κατά. Αποχές το ίδιο απορρίπτεται. 295 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 296 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 297 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 298 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 299 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 300 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 301 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 402 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 403 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 404 υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε. Πέρα στις οφορίες. 29 υπέρ, 28 κατά εγκρίνεται. 305 υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε και τη 305 ηλεκτρονικά. Άλλοι τρει να ψηφίσουν πέρα της ψηφοφορία. 24 υπέρ, 33 κατά, απορρίφθηκε. 306 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεν ψηφίζουν με τον ίδιο τρόπο οι μεγάλες ομάδες, οπότε είναι δύσκολο. 306 λοιπόν, πέρας. 23 υπέρ, 31 κατά απορρίφθηκε. 307 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 308 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 309 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 310 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. 310. Πέρας της ψηφοφορίας. 29-29 είναι το αποτέλεσμα. Αλλά η κυρία Πύρη ψηφίζει υπέρ, οπότε εγκρίνεται. 311 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 312 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 313 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 23 υπέρ 34 κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «320 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 321 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 323 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Λίγοι ακόμα. 23 υπέρ 34 κατά. 322 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61-325 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 324 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 326 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 326, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες, 33 υπέρ, 22 κατά. 327 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 328 υπέρ, 328, 328 υπέρ, κατά. Αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Πέρας της φοφορίας. 24 υπέρ, 33 κατά. 329 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 330 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 331 υπέρ και 332 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 333 υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 333 ψηφίστε παρακαλώ πέρας. 30-27. Εγκρίθηκε. 334 τώρα. Μάλλον όχι. Καταπίπτει. Πάμε στην 62-335. Υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, 337 λέει ο πρόεδρο. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 338 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63-339 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 340 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 340. Ψηφίστε παρακαλώ. 340. Πέρας της ψηφοφορίας. 25-28. Απορρίφθηκε. 341. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε και για αυτήν. 341. Thank you. Ευχαριστώ. 25-32 απορρίφθηκε. 3-4-2 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 343 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 343. 343 we are voting. 343 ηλεκτρονικά. in favor. 33 υπέρ 26 εναντίον εγκρίθηκε. 344 υπέρ. 344. Σηκώνετε τα χέρια παρακαλώ. Κατά. Απόχες. Θα λέγα εγκρίθηκε. 345 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίφθηκε. 346 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 347 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 351 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 352 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 353 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 65 354 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν 355 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε αλλά θα ελέγξουμε 355 ηλεκτρονικά άρχεται πέρας Απορρίφθηκε. 34 εναντίον, 23 υπέρ. Απορρίφθηκε. Ποια είναι τώρα? 356 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίφθηκε. 357 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίφθηκε. 358 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίφθηκε. 359 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 300 ποια είναι 300 α 67 361 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 362 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πως είπατε Ψηφίζαμε την 362, μόλις την ψηφίσαμε, εγκρίθηκε. Περνάμε στη συμβαστική 15, υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίθηκε. 365, υπέρ, κατά, απόχες. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 365 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε 29 υπέρ 28 εναντίον λοιπόν 366 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 367 συγγνώμη καταπίπτει αυτή 368 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 70, 370, 371 υπέρ αυτών. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. 372 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Η τροπολογία 72 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίφθηκε. 73 υπέρ. Διαμαρτυρία. Για ποια λέτε. Όχι δεν θα ελέγξουμε. Όχι. Πάμε στην 73 υπέρ. 73 υπέρ. Δεν θα ελέγξουμε την 72. Τέρμα. Αν θέλετε να καθίσετε δίπλα μου, εντάξει, ελάτε να ελέγξετε. Ήταν σαφές το αποτέλεσμα. 73 υπέρ. 73 υπέρ. Πολύ καλά. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 77 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 77 άρχεται πέρας απορρίφθηκε 23 υπέρ 33 εναντίον απορρίφθηκε συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 3 και 85 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 4 υπέρ δεν θα ελέγξουμε επειδή ήταν σαφέστατο το αποτέλεσμα. Πώς είπατε Γνωρίζω ότι δεν μπορείτε να δείτε τα χέρια ψυχώνων, εγώ τα βλέπω όμως. 86 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Η 6 και η 89 υπέρ αυτών. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 90 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 8 και 91 υπέρ αυτών κατά αποχές θα ελέγξουμε 8 και 91 άρχεται πέρας απορρίφθηκαν 35 εναντίον 92 τώρα υπέρ κατά κατά παρακαλώ αποχές θα ελέγξουμε. 92, δεν ήταν σαφέ το αποτέλεσμα. 92 ηλεκτρονικά άρχεται. Πέρας. 36 υπέρ, 20 εναντίον, εγκρίθηκε. 9. Η 93 ε, υπέρ της 93 κατά απόχες απορρίφθηκε. Συμβαστική 3 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 97 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 98 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 98 άρχεται πέρας εγκρίθηκε 32 υπέρ 26 εναντίον εγκρίθηκε 99 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Τελική ψηφοφορία τώρα όπως τροποποιήθηκε το κείμενο ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Tough vote. Παρακαλώ καθίστε. Ε, όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, να αποχωρήσετε. Οι άλλοι να καθίσουν γιατί έχουμε τον εκπρόσωπο της Βοσνίας τώρα παρακαλώ. Could you please take your seats and those who want to have a chat, they can either... Είστε και όσοι θέλουν ε, να παραμείνουν ή όσοι δεν θέλουν να αποχωρήσουν γιατί πάμε στο 5, σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης και είναι η ανταλλαγή απόψεων αυτό το σημείο με τον πρόεδρο του Συμβουλίου τον Υπουργό της Βοσνίας Εζεγοβίνης Πρωθυπουργό Ντένις Βίσντιτς. Καλώς ε, ήρθατε, καλημέρα σας, ε, σας χαιρετίζουμε, σας διαβιβάζουμε τις πιο θερμές μας, ε, τα πιο θερμά καλωσορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Επίσης θα ήθελα να χαιρετήσω τον εκπρόσωπο της <clears throat> Βοσνίας Εζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέσβυρα, Λίδια, Λίδια Είναι χαρά που σας έχουμε κύριε Βίστη στο Κοινοβούλιο. Εδώ και κάποιους μήνες ε, η ζήτησε η Βοσνία να είναι υποψήφια προσένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποψήφια προσένταξη χώρα και παραμένουν κάποιες μέρες ακόμα ώστε η αντιπροσωπεία της δικής μας Επιτροπής με επίσκεψη στο Μόσταρ και στη Βοσνία να γνωρίσει από πρώτο χέρι τις μεταρρυθμίσεις στη Βοσνία Ζεγοβίνη και πώς εσείς αντιμετωπίζετε τις δεσμεύσεις που είχατε αναλάβει και είχατε προσυπογράψει. Επίσης από την άλλη πλευρά το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε μια απόφαση ώστε να συστήσει στην Επιτροπή τη σύνταξη μιας έκθεσης σύνταξη έκθεση για την υποψηφιότητα τη Βοσνία Ερζεγοβίνη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια απόφαση πάρα πολύ ευαίσθητη και χρειάζεται η υποστήριξη των κρατών μελών. Ελπίζω να εγκριθεί. Ελπίζω να εγκριθεί κατά τη διάρκεια της Ολλανδική Προεδρίας. Αν όχι, υπό την ακόλουθη Προεδρία, υπό την Σλοβακική δηλαδή Προεδρία. Αναμένουμε να υπάρξει μια νέα δυναμική στο Συμβούλιο Υπουργών, μια νέα δυναμική μεταξύ των θεσμικών οργάνων Ελπίζουμε, ευελπιστούμε ότι η Βοσνία θα μπορέσει να υλοποιήσει, να συμπληρώσει αυτό το ερωτηματολόγιο επιτυχώ, που είναι η μεγαλύτερη προσπάθεια που πρέπει να κάνει μια χώρα η οποία έχει την φιλοδοξία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση έχουμε και την εφαρμογή τη συμφωνία, σύνδεση και σταθεροποίηση που άρχισε να ισχύει πριν από περίπου ένα έτο. Έχουμε μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων που βρίσκεται υπό εξέλιξη και επίση έχουμε μια ολόκληρη σειρά συμφωνιών που έχουν προχωρήσει ε, πολύ σημαντικά. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για αυτά τα θέματα πιο εξειδικευμένα και να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες από αυτών. Επίσης έχουμε και τον μηχανισμό συντονισμού, τον μηχανισμό, συντονιστικό μηχανισμό για τον οποίο έχει γίνει πολλής λόγος κατά τα τελευταία έτη. Χωρίς αμφιβολία έχει πολύ μεγάλη σημασία για την καλή λειτουργία όλων των διαδικασιών. Σας δίνω τον λόγο τώρα, έχετε 15 λεπτά, λυπούμαστε για την καθυστέρηση που δημιουργεί αλλά είχαμε ψηφοφορίες που ήταν ε, επίμαχες και γι' αυτό είχαμε κάποια καθυστέρηση. Επιπλέον οι ευρωβουλευτές θα σας θέσουν σίγουρα κάποιες ερωτήσεις στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, για μένα είναι τιμή και μεγάλη ικανοποίηση που έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Για μένα αποτελεί μια στιγμή καμπής για την πορεία μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η Βοσνία και η Ριζεγοβίνη είναι απολύτω αφοσιωμένη στην ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει ότι αποτελεί την ε, πρώτη μας προτεραιότητα όσον αφορά την εξωτερική μας πολιτική. Ξέρουμε ότι οι στόχοι είναι πολύ εσωτερική, εξωτερική, υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει τρομοκρατική απειλή που λαμβάνει όλο και περισσότερο παγκόσμιες διαστάσεις. Για μας λοιπόν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από την ε, ευρωατλαντική μας ε, ολοκλήρωση. Αυτό το οποίο είναι ουσιώδες για μας είναι το χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα φτάσουμε στους στόχους μας. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί κινητήριο δύναμη για τη δημοκρατία, για την πολιτική, για ε, την δικαιοσύνη, για τις υποδομές, για την ενέργεια. Όλα αυτά είναι αναγκαία για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Συνεπώ, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προποθέτει γενική πρόοδο στη χώρα μα. Θέλω λοιπόν να επαναλάβω για άλλη μια φορά κάτι το οποίο έχω πει πολλές φορές μέχρι σήμερα. Ότι δηλαδή ο ευρωπαϊκός δρόμος για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά δεν έχουμε άλλη αναλλακτική. Κυρίες και κύριοι. Μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας, Τώρα υπάρχει μια νέα όθηση και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Υπάρχει η πρωτοβουλία αυτή, η αγγλογερμανική, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ. Το Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο εκπροσωπώ, μου ζήτησε να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία αυτή. Έχουμε δει μέχρι τώρα ότι χάρη στην αλλαγή των προτεραιοτήτων ελευθερώθηκε και πάλι για μας ο δρόμος προς την Ένωση. Θέλουμε να εφαρμόσουμε τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις εκείνες οι οποίες θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών μας. Είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο το οποίο μας βοηθάει να ζούμε καλύτερα. Επίσης βλέπουμε ότι έχει ανανεωθεί και η πολιτική βούληση. Εμείς ανταποκριθήκαμε στο στόχο αυτό με πολιτική βούληση, με αποφασιστικότητα από πλευρά όλων των ηγετών στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το Σεβούλιο Υπουργών, το Κοινοβούλιο, όλα τα κυβερνητικά επίπεδα έδειξαν τη βούληση αυτή. Και είμαστε πεπισμένοι ότι ο μόνος δρόμος είναι ο ευρωπαϊκός. Επίσης, τελευταία σε όλα τα επίπεδα, κάναμε τεράστιες προσπάθειες για να ε, καλύψουμε τις, να συμμορφωθούμε προς τις προϋποθέσεις οι οποίε ε, τίθενται στο δρόμο μας για την Ευρώπη. Ο δρόμος αυτός είναι δύσκολος γιατί για να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις αυτό κοστίζει πολύ. Πρέπει να αλλάξουν οτροπίες για να το πετύχουμε. Όμως επειδή ακριβώς είχαμε τους στόχους αυτούς γι' αυτό καταφέραμε να βάλουμε προτεραιότητες και να προχωρήσουμε στο δρόμο αυτό που θα οδηγήσει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα λοιπόν και όλες οι αρχές έχουν μπει σε αυτό το δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Συνεπώς, σε αυτή τη θητεία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή αναγέννηση, ένα, μια νέα προσέγγιση ευρωατλαντική με νέε μεταρρυθμίσει. Η Βοσνία και η Ζεγοβίνη, κυρίε και κύριοι, όπω γνωρίζετε, ήδη από το Φεβρουάριο που μα πέρασε, υπέβαλε την αίτησή τη για υποψηφιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ένα τεράστιο στόχο για μα, το δρόμο μα αυτόν τον Ευρωατλαντικό. Και αποτελεί και ένα νέο κεφάλαιο στι σχέσει μα. Οι αξίε στι οποίε βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η δημιουργία ίσων ευκαιριών είναι αρχέ πάνω στις οποίες βασίζεται η οικονομική μας ανάπτυξη, η σταθερότητα και η ευημερία. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη με την υποψηφιότητά της αυτή έδειξε ότι είναι αποφασισμένη να αποτελέσει μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Και γι' αυτό ακριβώς έχω την ελπίδα ότι οι προσπάθειές μας, οι προσπάθειες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και ο ενθουσιασμός που έχουμε επιδείξει μέχρι τώρα θα αναγνωριστούν. Και έτσι, πολύ σύντομα, θα αποφέρει και καρπούς και θα αντικατοπτρίζεται στην στήριξη που μας δίνετε εσείς για να συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Κύριος στόχος μας είναι το ορατηματολόγιο. Το καθεστώς αυτό υποψήφιας χώρας ίσως για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μόνο τους τύπους. Για μας όμως, για τη χώρα μου και για τους πολίτες μας όπου το 80% θέλει την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί στρατηγική σημασία βήμα προς τη σταθερότητα και την ε, οικονομική και κοινωνική ευημερία. Γι' αυτό και θέλω να σας ε, παρουσιάσω τα μέτρα τα οποία έχουμε εφαρμόσει πρόσφατα. Και θέλω να επαναλάβω ότι συνεχίζουμε τη δουλειά μας προκειμένου να τηρήσουμε όλες τις προϋποθέσεις, όλα τα κριτήρια τα οποία μένουν ακόμα να εκπληρωθούν. Πολύ σύντομα θα το πετύχουμε. Πρώτον λοιπόν, προχωρήσαμε στην προσαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης και μετά θα αναφερθώ και στον μηχανισμό συντονισμού. Επίσης, εδώ και καιρό εφαρμόζουμε και μία ατζέντα στόχων. Ήδη τον Ιούνιο που μας πέρασε, Κάναμε μεγάλα βήματα. Συμπεριλάβαμε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων στον κοινωνικό τομέα, τον οικονομικό και τον δικαστικό. Από το 2015 μέχρι το 2018 προβλέπεται οι μεταρρυθμίσεις αυτές. Και ήδη το 2015 παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Όλα αυτά τα μέτρα έχουν, δείχνουν ότι οι προσπάθειές μας είναι αξιόπιστες ότι εμεί στο Συμβούλιο Υπουργών λαμβάνουμε τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά, τα οποία ήδη εφαρμόζονται πάνω από το 50%. Οι μεταρρυθμίσει αυτές είναι πολύ σημαντικέ. Είναι πολύ σημαντικέ για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της Βοσνίας και Σεγοβίνη, για την πρόοδό της. Και όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν έναν και μόνο στόχο, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Και έχουν εγκριθεί όλες οι στρατηγικές που περιλαμβάνονται στην ατζέντα μας αυτή. Με πιο σημαντική τη στρατηγική για τον, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα. Αυτή είναι μια μεταρρύθμιση η οποία βασίζεται σε διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βοσνία Ριζακοβίνη. Η στρατηγική αυτή συνοδεύεται και με τη στρατηγική τη καταπολέμηση τη τρομοκρατία και του εξτρεμισμού. Περιλαμβάνεται επίση και η αντιμετώπιση της διαφθορά. Έχουν εγκριθεί νόμοι, πολύ σημαντικοί νόμοι, όπως ποινικό, όπως εκείνο για τι διασυνοριακέ σχέσεις και η νομοθεσία εκείνη η οποία ρυθμίζει τον ε, δημοσιονομικό και φορολογικό τομέα, όπω επίση και τα εργασιακά. Οι νόμοι αυτοί και οι μεταρρυθμίσει αυτέ έχουν εγκριθεί στα διάφορα καντόνια τη χώρα. Για παράδειγμα, ο νόμο εκείνο που αναφέρεται στα εργασιακά, που εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θέλω να επαναλάβω ότι οι μεταρρυθμίσει αυτέ, οι περσινέ του 2015, πέτυχαν οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράμετροι στη Βοσνία Αρζεγοβίνη, οι δείκτε, να έχουν βελτιωθεί. Και αυτή είναι μια τάση η οποία συνεχίζεται και φέτο. Πέρυσι είχαμε 2,1% ανάπτυξη στο ΕΠ μας και πετύχαμε επίσης να δημιουργήσουμε 18.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Η παραγωγή αυξήθηκε, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,9% και το εμπορικό μας ε, έλλειμμα μειώθηκε. Αυξήθηκαν οι τουρίστες στη χώρα. Έτσι είμαστε από τις 10 χώρες του κόσμου που είχαν αύξηση στον τουρισμό τους. Οι εξαγωγές μας επίσης αυξάνονται σε όλους τους οικονομικούς τομείς, στην ενέργεια, στη γεωργία και σε άλλους κλάδους. Κάτι το οποίο μας κάνει να καταλάβουμε ότι τα προϊόντα μας έχουν καλύτερη ποιότητα όσο περνάει ο καιρός και ότι αναγνωρίζονται και σε άλλα σημεία της Ευρώπης. Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών είναι κυρίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 72% του όγκου των συναλλαγών αυτών. Και πρέπει να ολοκληρώσουμε με την έγκριση του πρωτοκόλου όσον αφορά τη Συμφωνία Σταθεροποίησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αυτών για μας προϋποθέτει ένα πολύ σημαντικό έργο. είναι πολύ σημαντικό και για τον ιδιωτικό τομέα, για την προστασία των παραγωγών μας, αλλά και πολιτικά έχει μεγάλη σημασία. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η προσαρμογή αυτή είναι από τα δύο ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ε, απόφαση το κατά πόσο θα είναι υποψήφια χώρα η Βοσνία Ζαγοβίνη ή όχι. Οι διαπραγματευτικές ομάδες αυτή την εποχή προσπαθούν να καταλήξουν σε μια γρήγορη λύση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά ακριβώς αυτό το στοιχείο, το καθεστώς, την απόδοση δηλαδή του καθεστώτος υποψήφιας χώρας. Από εκεί και πέρα υπάρχει πεποίθηση σε εμά ότι θα καλύψουμε τις προϋποθέσεις και θα μπορέσουμε έτσι να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου υπάρχει και ο μηχανισμός συντονισμού. Αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα συνταγματικά επίπεδα στη Βοσνία. Πρέπει να βελτιώσουμε την λειτουργία του. Γι' αυτό και πολλές φορές με με τους προέδρους της ομοσπονδιας Κροατομουσουλμανικής και με τον πρόεδρο επίσης της Σέρψκα. Και αυτό προκειμένου να ακούσω τις δικές τους προτάσεις, να τις λάβω υπόψη μου και να τις συμπεριλάβω στο οριστικό έγγραφο συντονισμού. Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο ήδη και πιστεύουμε ότι αυτός ο συντονιστικός ο μηχανισμός θα μπορέσει να συμπεριληφθεί στην γενικότερη δυναμική που θα μας βοηθήσει να συμπληρώσουμε το ερωτηματολόγιο. Όπως σας είπα, η πορεία μας προς την Ευρώπη είναι η προτεραιότητά μας και γι' αυτό και κάνουμε συνεχώς προσπάθειες για να το πετύχουμε. Βελτιώνουμε το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την οικονομική ευημερία στην περιοχή, την περιφερειακή συνεργασία και επίσης το πρόγραμμα δράσης, την αργοποίηση του προγράμματος δράσης για την ολοκλήρωση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας για να πετύχουμε μια Βοσνία και Ζεγοβίνη σταθερή και ευημερούσα. Έχουμε πολλούς στόχους μπροστά μας, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε με προσπάθεια, ώστε να πετύχουμε πρόοδο σε όλους τους τομείς που ανέφερα μέχρι τώρα. Θα δώσουμε αγώνα χωρίς να σταματήσουμε, άοπνα για να καταπολεμηθούν οι οργανώσεις οι τρομοκρατικές και εγκληματικές. Αυξήσαμε τον προϋπολογισμό μας των εθνικών υπηρεσιών που έχουν ως στόχο τους την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας και εξίσου από την άλλη πλευρά στρεφόμαστε στο να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο για όλες αυτές τις δράσεις. Επίσης, χάρη στις τελευταίες πρόσφατες προσπάθειες που κατεβλήθησαν σε αυτόν τον τομέα, μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε στη σωστή πορεία. Πάλι, από την άλλη πλευρά, ήταν φρικτές, φρικτά τα τελευταία πλήγματα στην Κωνσταντινούπολη, στο Λίβανο, στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών παγκόσμια και αυτό είναι υποχρέωσή μας, όλων μας. Γι' αυτό καταδικάζουμε τις τρομοκρατικές δραστηριότητες και τις θεωρούμε μία από τις μείζονες απειλές κατά της παγκόσμιας ειρήνης και γι' αυτό διπλασιάσαμε τις προσπάθειές μας για να ενισχύσουμε τις δομές και υποδομές μας για να επιτραπεί να διεξαχθεί ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας με επιτυχία. Επίσης ζητήσαμε από τις θρησκευτικέ κοινότητες να μας βοηθήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Η προσπάθεια αυτή είναι προτεραιότητα για μας. Πρέπει να έχουμε σχέσεις ιδιαίτερα θετικές με τους γείτονές μας. Αυτό είναι άλλος κύριος στόχος της εξωτερικής μας πολιτικής, διότι η ανάπτυξη της πολιτικής γειτονίας έχει θεμελιώδη ρόλο για την ε, οικονομική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα όλη της περιοχής μας, της περιφέρειάς μας. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε για την σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων και γι' αυτό εμείς και οι γείτονές μας έχουμε τις ευθύνες να αναπτύξουμε φιλικές και ειρηνικές σχέσεις μεταξύ γειτόνων. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά ότι πέρυσι έγιναν βήματα πως ε, μια σημαντική πρόοδο για να βελτιωθούν οι σχέσεις μας, ε, οι γειτονικές μας σχέσεις, κυρίως με τους πιο κοντινούς μας γείτονες. Για πρώτη φορά, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, συνήθαν οι εκπρόσωποι της σερβικής κυβέρνησης και της βοσνιακής κυβέρνησης. Και το ίδιο σχεδιάζουμε να πράξουμε και με τους εκπροσώπους της Κροατίας και τους δικούς μας. Σχεδιάζουμε και συντονίζουμε έτσι την προσπάθειά μας να προσχωρήσουμε, να ενταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατά τους επόμενους μήνες επίσης θα συνέλθουμε με εκπροσώπους από το Μαυροβούνιο, με τους οποίους επίσης συνεργαζόμαστε επιτυχώς. Και πράγματι υπογράψαμε επίσης από την άλλη πλευρά μια συμφωνία για τον καθορισμό των συνόρων των χωρών μας. Έτσι λοιπόν όπως και πέρυσι το 2015 στέφθηκε με επιτυχία το εγχείρημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αμφιβολία έχει θεμελιώδη ρόλο στο να μας υποστηρίξει σε αυτή την περιφερειακή πρωτοβουλία και προσέγγιση με συγκεκριμένα εξειδικευμένα μέτρα. Μεταξύ αυτών της διαδικασίας του Βερολίνου που δεν έχει μόνο πολιτική συνιστόσα αλλά και συνιστόσα για τις υποδομές και τα ενεργειακά θέματα. Για τη διασύνδεση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επίσης μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας μεταξύ των Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γιατί, διότι η διαδικασία του Βερολίνου ήταν κινητήρια δύναμη και μηχανή για να προαχθούν τα Δυτικά Βαλκάνια προς αυτή την κατεύθυνση. Πολλές φορές τα Δυτικά Βαλκάνια στις, στην Ευρώπη βρίσκονται σε ένα δεύτερο επίπεδο. Γι' αυτό ευκαιρίες όπως η σημερινή που συνερχόμαστε και συζητάμε δίνουν την προοπτική να ε, παραμείνει ανοιχτή η θύρα με τη διαδικασία του Βερολίνου και την Ευρωπαϊκή ημερήσια διάταξη το θεμα, θεματολόγιο για τη συνεργασία που έχουν θεμελιώδη ρόλο, ευελπιστούμε ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να δώσει ένα βήμα, να κάνει ένα βήμα προ τα εμπρό κατά τον Ιούλιο φέτο. Εκεί θα παρουσιάσουμε εμεί προγράμματα για τι μεταφορέ, τα ενεργειακά θέματα και το περιβάλλον. Όπως γνωρίζετε η Βοσνία Ζεγοβίνη κατά το 2015 πέρυσι προέδρευσε στο, ε, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και μέσα σε πλήρη κρίση, συγκυρία κρίση για το θέμα το, ζήτημα των προσφύγων μπορέσαμε έτσι να προσεγγίσουμε και να προαγάγουμε τα θέματα αυτά στην ευρωπαϊκή σκηνή. Για τον συντονισμό της ευρωπαϊκής καταπολέμησης της τρομοκρατίας για παράδειγμα που αφορά τους αλλοδαπούς μαχητές ε, στην ε, Μέση Ανατολή. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι και σε ετοιμότητα να ανταποκριθούμε στα όσα έχουμε δεσμευθεί να πράξουμε. Ολοκληρώνοντας θέλω να σας βεβαιώσω ότι η Βοσνία Ζεγοβίνη πλήρως ε, έχει αφιερώσει τις δυνάμεις της στην υλοποίηση των ε, αναγκαίων όρων για την ένταξη ε, αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας αυτά τα μέτρα τα οποία συζητούμε σήμερα συνεπάγονται μια προώθηση, μια νέα όθηση. Ευελπιστούμε ότι το Συμβούλιο θα έχει θετικά αποτελέσματα και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της θα λάβει θετικά υπόψη όλες μας τις προσπάθειες και όλα τα επιτέγματα μας πρόσφατα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την υλοποίηση και εκπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι δεν είναι κάποιο έπαθλο αυτό το ερωτηματολόγιο, αλλά είναι ένα μήνυμα υποστήριξης προς εμάς για την πορεία μας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς στη Βοσνία Ζεγοβίνη έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως τη σπουδαιότητα αυτού του εγχειρήματος και γι' αυτό έχουμε ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζουμε τις απαντήσεις μας σε αυτό το ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να δραχθώ τις ευκαιρίες για να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω για το σεβασμό σεβασμό που μας δώσατε σε σχέση με το ψήφισμά σας και την υποστήριξη που μας προσφέρατε στην πορεία μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ επίσης και για αυτό το ψήφισμα χωρίς αμφιβολία θα έχει μεγάλη σπουδαιότητα για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί με θετικό τρόπο να στεφθεί με επιτυχία η υποψηφιότητα της χώρας μας. Μας βοηθά σημαντικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη πλευρά εμείς είμαστε εκείνοι που είμαστε κύρια υπεύθυνοι. Χωρίς αυτή την υποστήριξή σας δεν θα είναι δυνατό βέβαια να ε, υλοποιηθούν όλα αυτά. Ευελπιστούμε ότι όλα αυτά θα μπορέσουν να στεφθούν με επιτυχία στο εγχείρημά μας. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να σας προσφωνήσω σήμερα. Η σχέση Όπω μας όπως αυτές οι σημερινή, η σημερινή μας συνάντηση είναι πολύ σημαντικές. Με τακτό χαρακτήρα σε συχνό, ε, συχνά να συναντώμεθα είναι πολύ σημαντικό. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε και έχετε πραγματικά πολύ μεγάλη πείρα πολιτική και επιπλέον είσαστε ο αρχιτέκτονας ε, ο οποίος εμπνεύστηκε και οικοδόμησε, δόμησε αυτή την προοπτική για την ευρωπαϊκή προσχώρηση, προσέγγιση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι ευρωβουλευτές κατέδειξαν και εκείνη τη δέσμευσή τους και την υποστήριξή τους προς τη Βοσνία Εζεγοβίνη από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευελπιστούμε ότι η δυναμική αυτή της Βοσνίας θα μπορέσει να επιταχυνθεί και πιο γοργά θα προχωρήσουμε από ό,τι στο παρελθόν και είμαστε έτσι πρωτοπόροι στις μεταρρυθμίσεις. Έξι συνάδελφοι ζήτησαν τον λόγο. Και αληθεύει βέβαια ότι έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο που προβλεπόταν για τη συνεδρίασή μας. 90 λοιπόν δευτερόλεπτα, 1,5 λεπτό κάθε ένας από όσους θα παρέμβουν. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε και να ξανασυζητήσουμε την Τετάρτη και την Πέμπτη στο Σαράγιο με τον κύριο Σφίτζης. Πρώτος ο εισηγητής κύριος Πρέντα και μετά η πρόεδρος της αντιπροσωπείας, ο, ο κύριος Πίτολα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ορίζω και εγώ εδώ τον ε, Πρωθυπουργό. Εδώ είσαστε μεταξύ φίλων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Εξάλλου ξέρουμε και τη συζήτηση που έγινε εδώ ε, για το ψήφισμα και την ψηφοφορία που ήταν ε, μια μεγάλη στήριξη προς τη χώρα σας. Θέλω να σας ευχαρώ όλους ιδιαίτερος για το θάρρος που έχετε επιδείξει μέχρι τώρα και να σας ανθαρρύνουμε. Θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε να λύσετε πολύ γρήγορα τα τρία ζητήματα τα οποία θα διευκολύνουν να επιτευχθεί στο Συμβούλιο Συνένεση όσον αφορά την απόδοση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας. Το είπατε κι εσείς και αναφερθήκατε σε αυτά τα τρία ζητήματα που είναι η εφαρμογή της ατζέντας με τις μεταρρυθμίσεις, ο μηχανισμός συντονισμού και η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Δεν χρειάζεται να επιμείνω εγώ περισσότερο. Συγχρόνως ελπίζω ότι θα πετύχετε τους στόχους που θέσατε, δηλαδή μέσα στο 2017 να πετύχετε την απόδοση του καθεστώτος αυτού υποψήφια χώρας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι. Για την ε, λεπτή αυτή υπόθεση, επειδή οι τοπικές εκλογές συγκλήθηκαν πριν από μία εβδομάδα από την ε, Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για όλη τη χώρα πλην της πόλης του Μοστάρ. Είναι μια κατάσταση που μας απασχολεί και θέλω να ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε και πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ευχαριστούμε τον Ίνος Βόλικα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ για όλα αυτά που κάνετε και αξίζετε συγχαρητήρια. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Το Νοέμβριο του 2014 ε, παρουσιάστηκε η νέα ε, προσχώρηση. Δεν ξέρω μετά από τόσο καιρό αν μπορούμε να μιλήσουμε για νέα προσέγγιση η οποία προκύπτει από τα πρώτα βήματα που προϋπήρξαν. Τώρα, σας ρωτώ ως πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών, πιστεύετε ότι μετά από 1,5 χρόνο η Βοσνία Ερζεγοβίνη αποτελεί μια ενιαία μακροοικονομική οντότητα, γιατί δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν ακόμα να γίνουν σημαντικές στρατηγικές και να εφαρμοστούν στον τομέα της ενέργειας και να ισχύσουν σε όλη την επικράτεια. Δεύτερον, ε, παρακολουθώ και το βοσνιακό τύπο βεβαίως και έχω την εντύπωση ότι η ανεργία των νέων είναι πάρα πολύ υψηλή. Εσείς ε, είπατε βέβαια ότι ε, αυτό το φαινόμενο το πρέπει να το καταπολεμήσετε σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα ως προτεραιότητα. Αλλά αυτή τη στιγμή υφίστανται διακρίσεις οι νέοι. Λέτε ότι θα έπρεπε να ε, μπορούν να συμμετέχουν στην οικονομική ανάπτυξη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Είναι δυνατόν με διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα να προβείτε σε συμφωνίες και να συνεργαστείτε μαζί τους για να καταπολεμήσετε ιδιαίτερα την υψηλή ανεργία των νέων στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, γιατί εκείνη είναι η παραγωγικότερη ηλικιακή ομάδα και μπορεί να αλλάξει και την κοινωνική δομή της χώρας. Ευχαριστώ ο κύριος Ράντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τη Βοσνία Ζεγοβίνη για όλα τα θετικά βήματα στα οποία προχώρησε και για την προοπτική της χώρας ε, να προσχωρήσει στην Ένωση. Βέβαια, έχετε να αντιμετωπίσετε μπροστά σας πολλά περίπλοκα θέματα ε, στα πλαίσια των υψηλών προτύπων που έχετε θέσει. Αναφέρατε το, την αύξηση του ΑΕΠ, τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 9%, ε, αύξηση των εξαγωγών, ε, του αγαθάριστου εθνικού προϊόντος. Όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία. Αυτή είναι, αυτές είναι οι προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν την ε, Βοσνία Ερζεγοβίνη στις δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Μια ερώτηση για την οικονομική ανάπτυξη. Πού στηρίζεται και πόσο σταθερή είναι και σε ποιο βαθμό μπορούμε να περιμένουμε ότι αυτό το θετικό πρόσημο της οικονομικής ανάκαμψης θα συνεχιστεί στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ε, ευχαριστώ τον κύριο Ράζο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω κάτι για κάτι που μας απασχολεί πολύ. Αυτή η διεκδίκηση των κρατών για μέρος η σύνολο της Βοσνίας. Ο κύριος Χωσάπεφιτς επίσης έκανε κάποιες δηλώσεις που μας ε, ανησυχούν πολύ γιατί μιλάει για το δοξασμένο παρελθόν το φασιστικό της Κροατίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση από πλευράς της Βοσνίας της Εγωβίνης. Πιστεύετε ότι αποτελεί μια απειλή από πλευράς της Κροατίας. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Παλμούιτα, νομίζω ότι υπερβάλλεται και ρωτάτε κάτι που δεν έχει καμιά σχέση με την επίσκεψη του κ. Βίστης. Δεν θα σας απαντήσω δημόσια εδώ, αλλά μεταγενέστε ιστερότερα θα, θα τοποθετηθώ. Έχει στη συνέχεια τον λόγο από πλευρά μα Σούιτσα, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι σχέσει με τη Βοσνία Ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με τη δήλωση του συναδέλφου Κόουσο, που κάνει λόγο για κροατικά θέματα που δεν έχουν καμιά σχέση με τη Βοσνία Εζεγοβίνη. Όπω είπε ο Αντιπρόεδρο, ελπίζω ότι αυτό μεταγενέστερα θα μπορέσει να αποσαφινιστεί. Συγχαρητήρια κύριε Σβητζήση για την εξαιρετική προσφώνησή σα ε, προ τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Η ταχύτητα της ολοκλήρωσης καθορίζει την ε, θετική έκβαση όλων αυτών και το ακούσαμε, γνωρίζουμε, ακούσαμε όλα τα στοιχεία, γνωρίζουμε τον ευάλωτο, ευαίσθητο χαρακτήρα όλων αυτών και για την βιομηχανία, αλλά τώρα για την ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, αυτά μας εξέπληξαν με θετικό τρόπο, πρέπει να πω. Θα ήθελα να μας απαντήσετε σε τι βασίζεται αυτή η οικονομική ανάπτυξη που είναι θεμελιώδους χαρακτήρα και είναι προτεραιότητα όπως είπατε. Είναι σαφές ότι οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει τώρα πλέον σε τι οφείλεται λοιπόν αυτή η κατάσταση. Για να μην επαναλάβω αυτά τα οποία γνωρίζουμε ήδη, θα ήθελα να θέσω άλλη ερώτηση. Αφορά την Ρεπούμπλικα Σέρψκα, τη Σερβική Δημοκρατία στην περιοχή σας. Είπατε ότι συνεργάζεστε με πολύ θετικό τρόπο σε όλα τα επίπεδα με τις αρχές της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Κάνατε λόγο επίσης για την ολοκλήρωση πολιτική της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και σε σχέση και με την Προεδρία της Ρεπούμπλικα Σέρψκα. Θα ήθελα να γνωρίζω αν η Ρεπούμπλικα Σέρβσκα θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα προσφέρει κάποια προοπτική ή θα αφαιρέσει κάποια προοπτική σε αυτές. Ευχαριστώ Ντουμπράφκα. Στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο συνάδελφος Καν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να πω ότι χαίρομαι που σας βλέπω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και εμείς οι σοσιαλιστές χαιρόμεθα διότι υπευλήθη η αίτηση για υποψήφια χώρα από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ στην πρόοδο που, που αναφέρατε κι εσείς. Θα είχα πολλές ερωτήσεις, αλλά περιορίζομαι σε μια ερώτηση που αναφέρθηκε και από του συναδέλφους. Έχει να κάνει με την ε, ε, τοπική κυβέρνηση του Μόσταρ ε, το από το 2008 επί 8 χρόνια δηλαδή και ανησυχούμε γι' αυτό δεν έχουν γίνει εκλογές Δηλαδή στερούνται ε, ένα θεμελιώδες δικαίωμα, δικαίωμα οι κάτοικοι εκεί. Επίσης, κατανοώ ότι μια πιθανή λύση για το πρόβλημα είναι να δημιουργηθούν δύο δήμοι για τη Βοσνία και την Κροατία. Αυτό με ανησυχεί βαθύτατα γιατί θα ήταν κάτι, πιστεύω, το οποίο θα μας πάει βήματα πίσω και όχι μπροστά θα ήθελα λοιπόν να μας το διευκρινίσετε αυτό και ποιους στόχους έχει η κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Βάλτο, Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, σας καλωσορίζω και εγώ θερμά. Είμαι πολύ ικανοποιημένος διότι ήρθατε σε μας με καλές ειδήσει τα δεδομένα και τα στοιχεία που μας δώσατε για την οικονομική ανάπτυξη είναι βεβαίως ε, καινούρια στοιχεία και πολύ θετικά. δεν υπάρχει μετάφραση. Υπάρχει κάποιο... Uh, Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την μετάφραση τη Σλοβενική φαίνεται. Όχι. Α. Να μιλήσω αγγλικά τότε. Θα μιλήσω αγγλικά. Χαίρομαι που υπάρχουν κάποια καλά νέα για την οικονομική ανάπτυξη. Και άλλα σημαντικά δεδομένα συναφή μας δώσατε. Θετικά όλα. Καλό είναι να έχουμε μια συζήτηση όπου δεν θα παρουσιάζεται ως πρόβλημα η Βοσνία Ερζεγοβίνη στα πλαίσια της ε, διεύρυνσης ε, ε, και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα. Η συνοχή σε ό,τι αφορά το διάλογο και την διαλλακτικότητα μεταξύ των εθνοτήτων είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ήταν στο παρελθόν, θα είναι και στο μέλλον. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό το στοιχείο λοιπόν στην κρατική σας μορφή πώς θα εξελιχθεί και να αναφέρω και τον κίνδυνο η Βοσνία να θεωρηθεί ως πιθανή πηγή Ισλαμικού εξτρεμισμού. Γιατί υπάρχουν ορισμένες τέτοιες πρακτικές και θα ήθελα τις διαβεβαιώσεις σας ότι έχετε αυτά τα φαινόμενα υπό έλεγχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βάιγκελ. Ε, κύριε Πρόεδρε, έχετε 6-7 λεπτά στη διάθεσή σας για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που έγιναν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Είμαι ευγνώμων και για την προσοχή που αποδίδεται στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις με τη σειρά. Καταρχήν, προς τους κυρίους Πρέντα και Καν, μπορώ να δώσω μια ενιαία απάντηση γιατί ήταν συναφείς οι ερωτήσεις και αφορούσαν τις εκλογές στο Μόσταρ που είναι ένα επίκαιρο θέμα στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ολόκληρη η πρόταση για τις εκλογές στο Μόσταρ ε, έτυχε επεξεργασίας από το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο των Υπουργών και εγώ δεν συμμετείχαμε καθόλου στη διαδικασία αυτή. Δεν υποβάλαμε προτάσεις εμείς για το Μόσταρ. Όμως θα ήθελα να αναφέρω κάποιες σαφείς αρχές που αποτελούν τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή για το Μόσταρ. Και είναι η εξή. Ο κύριος Χάνε μια ερώτηση. Το Μόσταρ δεν θα χωριστεί σε δύο εκλογικές μονάδες, ενότητες, ε, για τη Βοσνία και την Κροατία χωριστά. Δεν είναι αξιόπιστη πρόταση αυτή τώρα, καθόλου μάλιστα. Οι εκλογές στο Μόσταρ θα πρέπει να βασιστούν σε τρεις αρχές. Καταρχήν, δεν πρέπει να υπάρχει κυριαρχία μιας εθνοτικής ομάδας ε, πάνω σε άλλη. Δεν θα πρέπει να υπάρξει διαίρεση με βάση εθνοτικές ε, διαφορές, αναφέρομαι στις εκλογικές ενότητες, και θα πρέπει να ε, υπάρξει υποστήριξη στην ενιαία πόλη. Αυτές είναι αρχές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλες τις ενδεχόμενες προτάσεις. Και στα πλαίσια αυτών των αρχών θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα υπάρξει ένας δήμαρχος και δύο αντιδήμαρχοι, ίσως και τρεις, ε, γιατί είναι τρεις οι εθνότητες στο Μόσταρ και θα υπάρχει μια εναλλαγή, μια εκπεριτροπή στη Επίσης δεν υπάρχει φόβος να κάνουμε βήματα πίσω, να οπισθοχωρήσουμε στις λύσεις που επιδιώκουμε, αφού προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία ενοποιημένη πόλη, η οποία θα ε, λειτουργήσει και ως υπόδειγμα για την οργάνωση και άλλων πόλεων στη Βοσνία Ερζεγοβίνη με αυτόν τον τρόπο. Η δεύτερη ερώτηση από τον ε, αξιότιμο ε, συνάδελφο Τονίνη όπως είπατε, το Συμβούλιο Υπουργών ε, τώρα ε, υπάρχει εδώ και 14 μήνες. Η ανανεωμένη αυτή προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το θεματολόγιο των μεταρρυθμίσεων έπαιξε μεγάλο ρόλο τροποποιώντας, εναρμονίζοντας ε, την ε, μια αγορά στη χώρα. Οπότε η νομοθεσία σε επίπεδο οντοτήτων ε, και η, μεταρρυθμή, η νομοθεσία ε, έχει τώρα γίνει ενιαία. Δεν είναι δηλαδή κατακαιρματισμένη η αγορά. Όμως όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι χρειάζεται να γίνει ένα βήμα παραπέρα και να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση. Θα πρέπει να ε, παρουσιάσουμε εθνικές στρατηγικές και σχέδια τα οποία θα μας ε, βοηθήσουν να αναλάβουμε ε, πρωτοβουλίες ε, και να κάνουμε κοινά έργα. Έχουμε στρατηγική στον τομέα των μεταφορών, το περιβάλλον και την ενέργεια. Έχουμε επικεντρωθεί στην στρατηγική των μεταφορών. Τώρα που ελπίζομαι μέχρι τη Σύνοδο των ε, Παρισίων να ολοκληρωθεί. Ε, έχουμε δώσει όλη μας την ε, προσπάθεια εδώ. Αντικατοπτρίζονται εδώ οι προτεραιότητες της χώρας και μιλάμε τώρα εδώ για τις εσωτερικές και εξωτερικές μεταφορές. Θα συμπεριληφθούν προτεραιότητες και για τις διοντότητες σε εθνικό επίπεδο αλλά και στο κατώτερο επίπεδο της διακυβέρνησης ε, των καντονίων. Δεν θα σας κουράσω με Ξέρετε άλλωστε την κατάσταση, ε, ότι έχουμε ε, πάρα πολύ, ε, μια πάρα πολύ, ένα σημαντικό άξονα μεταφορών, ο οποίος θα παίξει κέριο ρόλο στην στρατηγική για τις μεταφορές, αφού θα λύσει πολλά προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής φύσης. Ε, επίσης, ε, κάναμε πρόοδο στην κατανόηση και αντιμετώπιση ε, της στρατηγικής μεταφορών σε σχέση με την οικονομία. Τώρα, για την ενεργεία των νέων είναι 24,5% αυτή είναι η γενική ανεργία. Η ανεργία των νέων φτάνει στο 60% και το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Τώρα, ε, ενδεχομένως ε, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους επιχειρηματίες για να προσλάβουν νέους ε, μέχρι 35 ετών. Στην Ομοσπονδία δεσμεύσαμε στα πλαίσια ενός προγράμματος κονδύλια για την απασχόληση ατόμων κάτω των 30 ετών. Έχουμε 7.000 νέους ανθρώπους που έχουν υποβάλει αιτήσει να συμμετέχουν και επίσης ε, με τη... έχουμε 750 ε, ε, έχουμε 750 εκατομμύρια δάνειο από από την τράπεζα για να επενδύσουμε σε τομείς ενδιαφέροντος στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Όμως ε, η πιστοτική αυτή γραμμή θα πρέπει να ε, αφιερωθεί ε, κυρίως στους νέους. Κάθε χρόνο δηλαδή το λιγότερο 50 εκατομμύρια δολάρια θα πρέπει να αφιερωθούν σε αυτό το τομέα. Για την οικονομική ανάπτυξη και αν είναι αυτή αξιόπιστη, η ερώτηση του κυρίου Ράντος είναι αξιόπιστη γιατί ε, αφορά ανάπτυξη που στηρίζεται στις εξαγωγές, στην, αύξηση, ε, στην καλύτερη ποιότητα των προϊόντων μας. Η παραγωγή ε, στηρίζεται σε εξειδικευμένο προσωπικό και ποιοτικές πρώτες Έχουμε την επεξεργασία ξυλίας που είναι πολύ σημαντική. Πέρσι ε, ξύγαμε ε, πάνω από 550 ε, εκατομμυρία και επίσης ε, είμαστε ε, από τις πρώτες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης εις ό,τι αφορά ε, την αυτοκινητοβιομηχανία, υφαντουργία για να μην μιλήσω για την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και πάλι λοιπόν είμαστε από τις χώρες που έχουν... επίσης έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση του τουρισμού αυξήθηκε ο τουρισμός κατά 25% και είχαμε και 20% ε, αύξηση των επισκεπτών ε, με βάση τα στοιχεία από τα ξενοδοχεία. Ε, Στην κυρία Σούισα, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και την υποστήριξή σας. Τώρα έχουμε μια ανανεωμένη προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη χώρα μας. Εμείς ε, έχουμε μια θέση και ε, το Κοινοβούλιο, η Κυβέρνηση, το Συμβούλιο των Υπουργών, η Αντιπολίτευση ε, συμφωνούν. Δεν έχει γίνει ποτέ διαφορετική δήλωση ούτε από την Ρεπούμπλικα Σέρψκα. Καμία δήλωση δεν υπάρχει που να είναι κατά της ένταξης. Βέβαια υπάρχουν ορισμένα εμπόδια σε αυτήν την ε, διαδικα... επιταχυμένη διαδικασία ε, προς την προσχώρηση. Αναλύουμε τον συντονιστικό μηχανισμό και είμαστε τώρα στο τελικό στάδιο. Σίγουρα η δέσμευση υπάρχει και αποφασιστικότητα βεβαίως. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς τα διαφορετικά κόμματα αντιλαμβάνονται την διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ε, θα πρέπει ε, να δούμε τρόπους ενδυνάμωσης του κράτους. Και προς τους ε, κυρίους Καν και Έντισον. Απάντησα στους προηγούμενους και τώρα για τον κύριο Βάγκερ. Στη Βοσνία Ζεγοβίνη υπάρχουν τρεις γλώσσες, επίσημες γλώσσες βοσνιακά, σερβικά, κροατικά. Σύμφωνα με το σύνταγμά μας. Αυτό πρέπει να το αναφέρουμε διαφοροποιούμενοι. Όσον αφορά τον εξτρεμισμό στη Βοσνία Ζεγοβίνη, καταβάλαμε πάρα πολλές προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είμαστε μία από τις λίγες χώρες που εισήγαγαν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ειδικέ διατάξεις στον ποινικό τους κώδικα, ποινικέ διατάξεις για να τιμωρούνται εκείνοι οι οποίοι επιστρέφουν και έχουν πολεμήσει σε τρίτες χώρες και είναι αλλοδαποί μαχητές. Επιπλέον η μουσουλμανική κοινότητα στη Βοσνία Ζεγοβίνη έκανε μια δήλωση σύμφωνα με την οποία αντιτίθεται πλήρως σε τέτοιου είδους πρακτικές. Τις καταδικάζει, όπως καταδικάζει και την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό. Και πράγματι, πρέπει να πούμε, η μουσουλμανική κοινότητα ήταν ο κύριος μηχανισμός και κινητήρας που μας επέτρεψε να τερματίσουμε, να αντιμετωπίσουμε τελεσίδικα αυτά τα ανεξέλεγκτα στοιχεία και να τα καταπολεμήσουμε. Η μουσουλμανική κοινότητα λοιπόν στη Βοσνία Ζεγοβίνη, υλοποιεί όλες τις διατάξεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί και βασιζόμαστε στη δέσμευση και εμπλοκή αυτής της κοινότητας που μας δίνει τη δυνατότητα πράγματι να συνεχίσουμε επιτυχώς την προσπάθειά μας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Και θα ήθελα να αποκαλέσω αυτή την περιοχή, περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η καταπολέμηση του εξτρεμισμού είναι βέβαια μια προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή μας ένταξη και προσχώρηση στην Ευρώπη. Ευελπιστούμε λοιπόν στις δεσμεύσεις των γειτονικών μας χωρών. Οι υπηρεσίες πληροφοριών μας επίσης ελέγχουν και επιτηρούν τα σύνορα και έχουμε διαπιστώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την καταπολέμηση τέτοιων ε, αυτού του είδους της μάστιγας όπως είναι η τρομοκρατία και ο εκτρεμισμός. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Σας ευχαριστούμε πολύ Πρόεδρε του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας απευθύνατε τον λόγο προσφωνώντας μας για τις μεταρρυθμίσεις στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είναι μεγάλη χαρά το ότι θα σας καναδούμε την επόμενη εβδομάδα στην αποστολή μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας άνοιξε την όρεξη για αυτή την αποστολή η επίσκεψή σας εδώ. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μεταξύ μας για τη σταθεροποίηση της χώρας σας. Εχθές στο Ντουμπρόμνικ υπήρξε μία σύνοδος ε, της ε, ομάδας των ε, κρατών του Ιωνίου Πελάγους και της Αδριατικής ώστε θα υπάρξει μια νέα προοπτική για αυτή τη συνεργασία. Σας ευχαριστούμε εσάς και την ομάδα σας. Και με αυτό ολοκληρώνουμε λοιπόν τη συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικών αλλά θα οδηγηθούμε αμέσω στην συνάντηση της αντιπροσωπείας για το Σαράγεβο στην, μετα... αποστολή μας αυτή πολύ σύντομα για μισό λεπτό για αυτή τη δέσμευση. στράτησε, το Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πω για αυτούς που θα πάνε στο Μόσταρ και στο Σαράγεβο. Έχετε πάρει την τεκμηρίωση ήδη που σας έχει αποσταλεί. Είναι ένα πολύ καλά διαθρωμένο πρόγραμμα. Θα φτάσετε είτε τρίτη απόγευμα βράδυ, που είναι το πιο ε, βολικό. Θα πάμε στο Μόσταρ. Το πρόγραμμα είναι νομίζω πάρα πολύ καλά διαθρωμένο. Η τεκμηρίωση έχει και στοιχεία και υλικά για όλη την ημερήσια διάταξη και εκδηλώσεις. Αν έχετε κάποιο συγκεκριμένο αίτημα να έρθετε σε επαφή με τον κύριο Μπάταρη ή και να αποστείλετε μήνυμα ώστε να σας βοηθήσουμε. Συμφωνείτε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε και ολοκληρώσαμε. Γεια σας.